Έχω ε, να σας κάνω την ανακοίνωση ότι η κυρία Μόνικα Μακοβέη εγκατέλειψε το ΕΛΚ και ε, προσχώρησε στο, στην ECR